να σας ευχαριστήσω η συγγήτρια Φωτίνκα για τα συμπεράσματά σας σε σχέση με την συμφωνία της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφγανιστάν. Ε, μετά από δεκαετίες πολέμου, το Αφγανιστάν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Πέρσι ήταν η πιο... Ε, Θανατερή χρονιά για τους πολίτες εκεί. Το 2018 θα μπορούσε να είναι το έτος της ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάστηκε πιο στενά ακόμα με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν για να συνοδεύσει τη χώρα αυτή την λεπτή στιγμή που περνάει στην ιστορία του. Αυτός είναι και ο στόχος μας στη στρατηγική μας που θέσαμε ήδη από το 2017 και στα συμπεράσματα επίσης του Συμβουλίου. Η συμφωνία αυτή λοιπόν αποτελεί το πρώτο νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μας με το Αφγανιστάν και απορρέει από μακρές διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Η συμφωνία τώρα εφαρμόζεται προσωρινά. Ήδη όμως έχουμε μια πολλά υποσχόμενη αρχή του διαρθρωμένου μας διαλόγου και της συνεργασίας μας. Έχαμε ήδη το 2018 δύο διμερείς συνεντήσεις όπου συζητήσαμε πολλά κομβικά ζητήματα για τα οποία συμφωνήσαμε με τους Αφγανούς φίλους. Μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θέματα ισότητα μεταξύ των δύο φίλων, χρηστή διακυβέρνηση, συνεργασία, εμπόριο, περιφερειακή συνεργασία. Για όλους αυτούς τους φακέλους, το Αφγανιστάν θέλει να προχωρήσει προς όφελος των πολιτών του. Και εμείς, οι Ευρωπαίοι, προσχεθήκαμε βοήθεια και στήριξη δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση που επικρατεί με τους Αφγανούς πρόσφυγες στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη να συνεργαστεί για μια ικανοποιητική και συνολική λύση προκειμένου να μπορέσουν συντεταγμένα και με ασφάλεια να επιστρέψουν οι Αφγανοί στη χώρα τους που τώρα ζουν στις γείτονες χώρες και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Μετανάστευση και τους Μετατοπισμένους. Στην έκθεσή σας, εσείς, ε, σκεγγραφείτε ρεαλιστικά την κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα εγώ να επεκταθώ λίγο περισσότερο στις τρέχουσες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την ειρήνη. Η κατάσταση επιτόπου παραμένει δύσκολη. Αυγανοί, αθώοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη σύγκρουση. Υπάρχουν όμως αρκετοί λόγοι για να αισιοδοξούμε και να έχουμε κάποια καλά νέα από τη χώρα. Ο πρόεδρος προσέφερε ερνευτικές συνομιλίες το Φεβράριο του 2018 με τους Ταλιμπάν, πριν δηλαδή από ένα χρόνο περίπου. Δημιούργησε έτσι μια καλή προϋπόθεση για την ειρήνη. Και από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι Ταλιμπάν πραγματεύονται για απόσυρση και για δεσμεύσεις. Ξέρετε ότι για να έχουμε μία ειρήνη διάρκειας χρειάζεται χρόνος. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίξει το Αφγανιστάν πριν και μετά την ειρηνευτική λύση προκειμένου η ειρήνη να είναι διαρκεία. Στον Εύρο που μας πέρασε, στην Υπουργική Διάσκεψη στη Γενέβη για το Αφγανιστάν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η ύπατη Εκπρόσωπο Μογκερίνη παρουσίασε πέντε σημεία και τα πρόσφερε στο Αφγανιστάν για το πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να στηρίξει την ειρήνη. Πρώτα απ' όλα, η ειρηνευτική διαδικασία να προχωρήσει με τη συμμετοχή όλων, χωρίς αποκλεισμού. Δεύτερον, να βοηθήσουμε στις μεταρρυθμίσεις, ακόμα και στον τομέα της ασφάλειας. Τρίτον, να βοηθήσουμε με την επανένταξη των παλιών μαχητών και των οικογενειών τους. Τέταρτον, να δράσουμε ως εγγύτης σε μια ερηνευτική συμφωνία. Και τέλος να ενισχύσουμε το εμπόριο και την ε, διασυνδεσιμότητα. Έκτοτε συνεργαζόμαστε με τους Αφγανούς εταίρους μας προκειμένου να καθορίσουμε καλύτερα πώς θα προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια. Έχουμε ξεκινήσει με έναν ειρηνευτικό μηχανισμό για να χτιστούν ικανότητες στη χώρα. Όπως είπε στη Γενέβη, είπατε εκπρόσωπος, οι Αφγανοί ζητούν να προχωρήσουν προς τα μπρος. Δεν υπάρχει περιθώριο να πάνε πίσω. Τους επόμενους μήνες λοιπόν θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να στηρίξουμε μια καλύτερη εκλογική διαδικασία για τις φετινές προεδρικές εκλογές στο Αφγανιστάν. Όπως σωστά λέτε και εσείς στην έκθεσή σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει μεγάλη χρηματοδότηση ως αναπτυξιακή βοήθεια. Στην διάσκεψη των Βρυξελών τον Οκτώβριο του 2016 για το Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη προσέφεραν 5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει αρχίσει να λειτουργεί η βοήθεια αυτή. Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι η αναπτυξιακή στήριξη στο Αφγανιστάν επικεντρώνεται κυρίως στην ειρήνη, στην οικοδόμηση του κράτους και στηρίζει το Αφγανιστάν περιφερειακά. Με άλλους αναπτυξιακούς εταίρους επίσης προσπαθούμε να βρούμε πώς θα προσαρμόσουμε τα αναπτυξιακά μας προγράμματα βάσει αυτού ακριβώς του σεναρίου. Προκειμένου να συμπεριλάβουμε μεταρρυθμίσεις, κοινωνική συνοχή σε κοινοτικό επίπεδο και διασυνοριακό εμπόριο και διασυνδεσιμότητα. Το Αφγανιστάν έχει μια μοναδική ευκαιρία τώρα για ειρήνη. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να βοηθήσουμε τους Αφγανούς να αποφεληθούν από την ευκαιρία αυτή και να την καταστήσουν μια περίοδο ειρήνης διαρκείας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα, κύριε Επίτροπε, συνεχίζουμε με τον κύριο Έγγελ. Ε, θα έπρεπε αυτός να πάρει το λόγο, όμως δεν τον βλέπω εδώ. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Λάγκε. Εκ Επιτροπής Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κάπως παράδοξη η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρέπει να εγκρίνουμε ε, μια συμφωνία η οποία έχει προσωρινά τεθεί σε ισχύ ε, ήδη εδώ και ένα χρόνο και που κατά την διαπραγμάτευση δεν υπήρχε καμία διαφάνεια. Κανονικά δεν είναι τρόπος αυτός να συμπεριφέρεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και δηλώνω απερίφραστα στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να τίθενται σε ισχύ συμφωνίες χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του αυτό το δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία αυτό. Έχουμε πει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ προτού δώσει τη συγκατάθεσή του, την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό το απευθύνω ως αίτημα στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Εμείς είμαστε το δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δικαίωμα να συμμετάσχουμε στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις και προτού τεθεί οποιαδήποτε συμφωνία σε ισχύ θα πρέπει να διαβουλεύεστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντρογεύσκη έχει το λόγο. του Europejskiego do jakiejkolwiek współpracy. Ta współpraca natomiast wkracza w tej chwili w decydującą fazę i na tym etapie ta zgoda jest Χρειάζεται συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αποφασιστική σημασία. Η έγκριση είναι πολύ σημαντική. Χαίρομαι που η Επιτροπή ΑΦΕΤ δέχτηκε και είδε με θετικό μάτι αυτή τη σύσταση Ξεκινά λοιπόν η πρώτη επισήμη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν. Μ' αρέσει όμως επίσης και η έκθεση που την θεωρώ ότι είναι πληρέστατη. Εμπεριέχει πολιτικές στρατηγικές πτυχές, αναφέρεται στο ρόλο των περιφερειακών φορέων, αναφέρεται σε θέματα πάπτω της ασφαλείας και της ε, ειρήνευσης στο Αφγανιστάν, αναφέρεται και στην ε, δημιουργία του κράτους, διότι το Αφγανιστάν είναι κράτος ε, που τελεί υπό οικοδόμηση. Αναφέρονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα που στα Αφγανιστάν παραβιάζονται πολύ συχνά. Αναφέρεται στην οικονομία, στην ανάπτυξη, αναφέρεται στο εμπόριο, αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή που είναι κλειδί, που είναι των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το Αφγανιστάν ε, ε, δεν είναι έτοιμο ακόμα να καλύψει τις ανάγκες των μεταναστών πηγαίνουν οι Αφγανοί στο Πακιστάν. Χρειάζεται μια συνεργασία και σε αυτό το μέτωπο και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πληρέστατη αυτή η έκθεση. Ο πρόεδρο λέει ευχαριστώ. Εν ονόματι τη ομάδα SND, ε, ο κύριο Φραντσούλικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Συμφωνία Συνεργασίας για Σύμπραξη και Ανάπτυξη επιβεβαιώνει την αφοσίωση στην στήριξη ε, της ανάπτυξης του Αφγανιστάν το 2014-2024 και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε βασικές ε, αλλαγές στη χώρα. Μάλλον 2019-2024. Παρά τη σημαντική πρόοδο που ετεύχθη, το Αφγανιστάν ακόμα αντιμετωπίζει ουσιαστικές προκλήσεις που χρειάζονται ε, μεγαλύτερη δύναμη, επί μεγαλύτερη διάρκεια για να πετύχουμε τους στόχους. Τονίζουμε ότι χρειάζεται επικοδομητικότος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που είναι συστατικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Η συμφωνία στόχο έχει να αναπτυχθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσης Αφγανιστάν σε ένα όλο και ευρύτερο φάσμα ευνοϊκών δομιών. Καταπολέμηση εξτεμισμού, τρομοκρατίας, κράτος δικαίου, βελτίωση ε, διακυβέρνησης, ειρήνη, ανάπτυξη, καταπολέμηση της οικονομικής ενίσχυσης των τρομοκρατών, ε, το ελευθερμπόριο ναρκωτικών καταπολεμηθεί, να προωθήσουμε ανάπτυξη πέθρου, κοινωνική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουμε από κοινού την πρόκληση αλλαγή του κλίματο. Το Αφγανιστάν θα πρέπει να συγκρατηθεί από το να προωθεί ε, δια εκπροσώπων μάχε στην περιοχή. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στη σταθερότητα στο Αφγανιστάν αντί να το υπονομεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο, ο κύριος ε, έχει το λόγο για την Άλντε. Κύριε Πίτροπε, συνάδελφε, καταρχά θέλω να ευχαριστήσω την Άννα Φωτίνκα για την ε, άριστη δουλειά τη ε, και την έκθεση αυτή που παρουσιάζεται σήμερα και που συζητούμε. Η Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκή Ένωση Αφγανιστάν φέρνει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αφγανιστάν σε ένα νέο ποιοτικό επίπεδο για την αμοιβαία εποφελή συνεργασία. Αναμφισβήτητα, το Αφγανιστάν έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο σε πάρα πολλούς τομείς, όπως σωστά αναφέρει Ανέφερε και η Άννα. Ωστόσο, ανησυχίε για την ασφάλεια, ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διαφθορά εξακολουθούν να υπάρχουν και θέτουν σε κίνδυνο τα επιτεύγματα μέχρι σήμερα. Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο στην ε, ιστορία του, καθώς αν δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μπορεί να πάνε χαμένες οι προσπάθειες που έχουν γίνει. Η συμμαχία που έχει ε, δημιουργηθεί ε, θα πρέπει να έχει πάντοτε την συμφωνία και τη συγκατάθεση όλων των συμμάχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσωλωμένη σε μια μακροπρόθεσμη σχέση συνεργασίας με, την, ε, με το Αφγανιστάν. Έπειτα λοιπόν από την Σύνοδο της Γενέβης για το Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χρηματοδοτικό πακέτο ε, ύψους 470 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχυθούν οι υποδομές, η δικαιοσύνη, το σύστημα υγείας και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μετανάστευσης και εκτοπισμού στο Αφγανιστάν. Ελπίζω λοιπόν η συμφωνία αυτή ε, θα εδράζεται σε μια περιφερειακή προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει τους γείτονες του Αφγανιστάν. Η διεθνής κοινότητα μπορούν να χαράξουν το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Πρώτο βήμα σε αυτή την πορεία της σταθερότητας θα είναι η ειρήνη. Η επίτευξη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των αντιμεχόμενων πλευρών στο Αφγανιστάν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω πραγματικά η διαδικασία κατά των διαπραγματεύσεων να συμπεριλάβουν την ε, κυβέρνηση του Αφγανιστάν με την πραγματική έννοια, συγκεκριμένα. Μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να θέτει σε υποαμφισβήτηση τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το αξίζουν οι πολίτες του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Λόζινγκ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό εκ μέρου της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Είναι θετικό όταν οι στόχοι συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωση και, ε, ε, και του Αφγανιστάν, όπως η καταπολέμηση τη φτώχεια, η ισότητα των φύλων, η επίτευξη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται ε, σε, ίδια προτεραιότητα. Όμως δεν είναι ότι δεν έχουμε εμπειρία ε, όσον αφορά νεοφιλελεύθερε μεταρρυθμίσει, τι οποίες εισάγει αυτή η συμφωνία. Ήδη από το 2003 η Δύση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εισήγαγε ε, και ξεκίνησε μια ριζική αναδιάρθρωση σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση του οικονομικού συστήματος της χώρας. Ωστόσο, εδώ και χρόνια διαπιστώνεται ότι τα μέτρα που υπαγορεύτηκαν στο Αφγανιστάν δεν έχουν βοηθήσει ούτε στο να βελτιωθεί η κατάσταση του λαού ούτε και της οικονομίας της χώρας. Η συμφωνία αυτή είναι καταστροφική για το λαό του Αφγανιστάν. Η προώθηση των ξένων επενδυτών του ιδιωτικού ταμείου και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας δεν θα βοηθήσει τη χώρα να σταθεί στα πόδια της, αλλά θα ε, διευρύνει, και αυτός είναι ο στόχος της, τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επίσης, η συμφωνία συμπεριλαμβάνει, και εδώ βάζω θαυμαστικό, εκ των προτέρων άτυπες συμφωνίες ε, επιστροφής με το κοινικό όνομα «Μαζί οδεύουμε μπροστά» που στην πραγματικότητα ε, στέλνει ανθρώπους πίσω στο Αφγανιστάν, δηλαδή στο θάνατο. Αυτή η πρακτική πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφορες αποστολές του ΟΙΕ που πάνε να προστατεύσουν ε, διάφορες μειονότητες, στις γυναίκες για παράδειγμα. Δυστυχώς όμως είναι αιματηρή η ιστορία. Δεν υπάρχει ειρήνη όσο υπάρχει αποκλεισμός. Τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, απόσυρση στρατευμάτων. Όλα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά γιατί ούτε η κοινωνία των πολιτών, ούτε οι γυναίκες, ούτε η νεολαία έχουν φωνή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για μια απειλή. Ο περισσότερος κόσμος, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι έφηβοι θα βρεθούν να καταπιέζονται με βαρβαρότητα. Πρόκειται για προδοσία. Όλο και περισσότερες επιθέσεις έχουμε από τους Ταλιμπάν εναντίον των στρατιωτικών στο Αφγανιστάν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δικιά της την πλευρά τι κάνει. Η συμφωνία αυτή δεν αξίζει το χαρτί πάνω στο οποίο γράφεται. Πρόκειται για οπισθοχώρηση του πολιτισμού. Αυτή η συμφωνία σύνδεση και συνεργασία δεν πρόκειται να βοηθήσει. Όλε οι ανθρωπιστικέ προσπάθειε οδηγούν σε θυσία των Αφγανών και των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν θα έχει βοηθήσει σε τίποτα όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τζίλ. Ξέρω ότι η συμφωνία αυτή υπάρχει και ότι σίγουρα θα ήταν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ενημερωθεί πιο έγκαιρα για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά κυρίως τις επενδύσεις και το εμπόριο. Όμως, παρόλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι η Ουάσιγκτον δεν πιέζει για στρατιωτικό ε, προβάδισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει πολιτική λύση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν. Έχω διάφορες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαπραγματευτές Λιμπάνωμένων Πολιών έχουν καταλήξει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο, το οποίο όμως δεν έχει κυκλοφορήσει Ποια είναι τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις μειονότητες ή τις γυναίκες στο Αφγανιστάν, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες για περισσότερη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο βίο. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν γίνεται αυτομάτια και ότι δεν θα έχουν πολιτικό ρόλο οι Ταλιμπάν. Έπειτα, δεν υπάρχει περιφερειακό πλαίσιο συμφωνίας. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε το Αφγανιστάν μπορεί να προχωρήσει πώς θα διασφαλίσουμε ότι στην περιφέρεια το Πακιστάν, η Ινδία και το Ιράν θα βοηθήσουν να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Πώς θα υπάρξει πρόσβαση και δική μας το διάλογο αυτό και στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Ward είναι η πρώτη. Mm. Τα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω εξακολουθούν να θεωρούν ότι το Αφγανιστάν είναι μια ασφαλή χώρα. Αυτό επιτρέπει να επιστρέψουν στη χώρα ανθρώπου που ήρθαν στην Ευρώπη για να ζητήσουν άσυλο πολύ συχνά ε, μέσω από πολύ επικίνδυνε διαδρομέ. Όμω η κατάσταση επιτόπιση των αφορά την ασφάλεια έχει επιδεινωθεί σοβαρά και οι Ταλιμπάν ελέγχουν σημαντικό κομμάτι τη επικράτεια. Είναι υποκριτικό και ανεύθυνο τα κράτη-μέλη μας να στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους πίσω σε μια χώρα όπου αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουν δίωξη, κυρίως εκείνοι που ήρθαν να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη αφού ήταν στόχος λόγω της συνεργασίας τους με τις δυτικέ δυνάμεις. Άλλο ανησυχητικό θέμα είναι ο παρόν αποκλεισμό γυναικών και νέων από συνομιλίε που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ταλιμπάν. Η συνάδελφό μου, Ιάννα Γκόμε, ε, μας ε, έθεσε υπό προσοχή μια σημαντική πρωτοβουλία. Μία ομάδα γυναικών από το Αφγανιστάν έκαναν απέθανα έκκληση για εκείνους που ξερούνται από τις συνομιλίες. Είναι σημαντικό να εισακουστούν οι φωνέ του για να οικοδομηθεί μια βιώσιμη Ευρώπη και να διαφυλαχθούν τα ε, δικαιώματα των γυναικών στη χώρα που τα κέρδισαν με σκληρού αγώνε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λαλάντας. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια συμφωνία έχει συναυθεί μεταξύ Ταλιμπάν και ΙΠΑ εδώ και μερικές ώρες στην Τόχα. Μέχρι χτε επιτέθησαν οι Ταλιμπάν σε, με 50, σε 50 στρατιώτε του Ταλιμπάν, 16 σκοτώθηκαν και 40 φυλακίστηκαν. 10 μέρε πριν, 40 στρατιώτε σκοτώθηκαν στου Ταλιμπάν στη νότια περιοχή τη χώρα και μπορώ να πλησιάσω τα διάφορα πρόσφατα παραδείγματα. Οι Ταλιμπάν αρνούνται πάντα να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν παρά τα επανειλημμένα αιτήματα τη κυβερνήσεω. Αυτοί πολλαπλασιάζουν τι επιθέσει κατά τη κυβερνήσεω και τελευταία, μόνο το 50% η κυβέρνηση ελέγχει τη χώρα. Λοιπόν, προγραμμάζεται μια πολιτική επιστροφή ε, των Ταλιμπάν στην εξουσία σε εθνικό επίπεδο βάσει αποδυναμωμένου εκτελεστικού. Αυτό είναι πρόβλημα για τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη των δικαιωμάτων και κυρίως των γυναικών. Η κοινωνία του Αφγανιστάν όλοι ανησυχεί που βλέπει εκ νέου να δημιουργείται ένα Ισλαμικό Εμμυράτ ε, στο Αφγανιστάν που σκοτώνει την ελευθερία, όπω γινόταν και δεκαετία του 90. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί λόγω αξιοπιστία τη να επιτρέψει να στηρίξει ένα τέτοιο δεχόμενο μετά από 20 χρόνια επενδύσεων στο Αφγανιστάν. Κύριε Επίτροπε, δεν μπορούμε να αφήσουμε του Αφγανού να ξαναπέσουν στι ίδιε μέρε ε, ε, που οδηγούν ε, τι διαδικασίε συνευτικέ και κυβερνούν εν ονόμα τη ειρήνη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Μιας και συζητάμε το Αφγανιστάν, το κράτος που ιστορικά ήταν πάντοτε αδύνατο να κυβερνηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει τη χώρα αυτή, ε, προσφέρει επενδύσεις, ε, οικοδόμηση κρατικών θεσμών, δημοκρατία, σύστημα υγείας. Τώρα από την άλλη πλευρά υπάρχουν η ΙΠΑ, η Ρωσία ε, και η Βρετανική Αυτοκρατορία που όλες απέτυχαν να επιβληθούν στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη ήπια δύναμή τη προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά τη συμφέροντα στο Αφγανιστάν. Εγώ νομίζω ότι για να ε, ωφεληθεί πραγματικά ο λαό του Αφγανιστάν θα πρέπει να υπάρξει ανοιχτό εμπόριο για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσω του εμπορίου να ζήσουν οικονομική ανάπτυξη και παιδεία. Οτιδήποτε άλλο είναι καταδεκασμένο να αποτύχει. Ευχαριστώ πολύ και τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Καστάλντο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, το Αφγανιστάν παρόλο που είναι κοντά στην ευαισθησία μας και κοντά στους πολίτες Ευρωπαίους ε, λόγω των πεσόντων που προέρχονται από τα κράτη-μέλη, του συμμάχου που θυσίασαν τη ζωή του στρατιώτε εκεί. Και σήμερα θα ήθελα αυτό να το επενθυμίσω. Τούτο λεχθέντο πιστεύω ότι το Αφγανιστάν, όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται μια συμφωνία που υποστηρίζει τον πολιτικό διμερή διάλογο για να παγιωθεί σταθερότητα στη χώρα, χωρί όμω να λησμονούμε και μάλιστα να θέτουμε στο επίκεντρο τα δικαιώματα των πολιτών, το κάτω δικαίου, τη μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση τη διαφθορά. Στα πλαίσια της Κεντρικής Ασίας που αλλάζει, η σταθερότητα του Αφγανιστάν είναι επωφελής για όλους, για όλους τους περιφερειακούς φορείς. Χωρίς συμμετοχή στο σπάθι του ΟΗΕ δεν θα είναι επαρκείς οι προσπάθειε και σίγουρα θα είναι πιο δύσκολες οι προσπάθειε. Πέρα από τη σταθερότητα, η συμφωνία έχει σαν λογική συνέπεια έναν έλεγχο των πόρων, σημαντικότατη πτυχή για μα, ώστε αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιούνται πραγματικά υπέρ των τοπικών πληθυσμών. Είναι δύσκολο ο δρόμο, αλλά αυτό είναι πρώτο θετικό βήμα και θα πρέπει να ανοίξουμε τι πόρτε, να κρατήσουμε ανοιχτέ για ελπίδα για ένα μέλλον για του πολίτε του Αφγανιστάν. Ε, Ευχαριστούμε. Εδώ η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την παρέμβαση του Επιτρόπου. Ο κύριος Μίμητσα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο χρήσιμη συζήτηση. Καταλήγω στο ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας με το Αφγανιστάν και γενικά με τι προσπάθειε της Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τη χώρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, σε αυτή τη στιγμή όπου όλο και μεγαλύτερη δέσμευση χρειάζεται συνολικά από τη διεθνή κοινότητα. Εμείς ε, θα αποζητούμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ε, διάλογο και τη συνεργασία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα η κυρία Φωτίγκα. Η συγκίτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η συμφωνία συνεργασίας, εταιρική σχέσης και ανάπτυξης είναι η πρώτη αυτού του είδους ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αφγανιστάν. Πρέπει να παραμείνει για την επόμενη δεκαετία και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε πλήρως προκειμένου να προσφέρουμε ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη, όπως επίσης ε, να φροντίσουμε η χώρα αυτή να είναι και κοινωνικά βιώσιμη. Είναι δύσκολο έργο. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες εισηγητές, όλους όσοι συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή, του συμβούλους της πολιτικής μου ομάδας, το προσωπικό της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και του δικούς μου βοηθούς. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πρόεδρος. Ευχαριστώ και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε στην ε, συζήτηση αυτή και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης Έκθεση Χουάν Φερνάντο Λόπε Αγγιλάρ, Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Μονακό, τη Ανδόρα και του Αγίου Μαρίνου. Πρώτο έχει τον λόγο ο εισηγητή. Παρακαλώ. Έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας, κύριε Αγγιλάρ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μίμητσα, είναι τιμή για μένα που παρεμβαίνω στην Ολομέλεια αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εισηγητή για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Συμφωνία σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το Πριγκιπάτο του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2014 το Συμβούλιο επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου των χωρών μελών να διαπραγματευτεί μια συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα σε αυτές τις μικρής ε, έκτασης ε, χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι εξέφρασε την ε, επιθυμία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε, να τοποθετηθούμε πριν λήξει η θητεία μας για την συμφωνία αυτή σύνδεσης. Και δεν θα μπορέσει, μην το γνώμε αυτό, να εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή σύνδεσης αν δεν δώσετε σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πάντα στις διεθνείς συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λόγο με την σύμφωνη γνώμη μας. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια μακρά ιστορία στην διαδικασία αυτή που θα ήθελα να την θυμίσω κάπως, μια που είμαι και καθηγητής ε, για τέτοια ζητήματα. Είχαμε διαπραγματεύσεις λοιπόν για τη συμφωνία αυτή σύνδεσης. Αυτό όμως που διαπίστωσα είναι ότι και οι ε, όμορες χώρες, η Γαλλία ας πούμε και η Ισπανία, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη συμφωνία σύνδεσης, γιατί είναι πολύ σημαντική η εταίρη. Και έτσι αυτές οι τρεις χώρες, παρόλο που γεωγραφικά έχουν πολύ μικρή έκταση, είναι ε, σημαντικές και ας έχουν και λίγο πληθυσμό. Βάσει του άρθρου 8 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουν δικαίωμα ευελιξίας και ρεαλισμού όταν ενσωματώνουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις τέσσερις ελευθερίες. Να υπάρχει νομική ασφάλεια, αλλά να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες των τριών αυτών χωρών όταν ενσωματώνουν το κοινοτικό κεκτημένο. Γιατί είναι σαφές ότι σε σχέση με την εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών σε μια τόσο μικρή γεωγραφικά ε, χώρα, προφανώς και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας και επαναδιαπραγμάτευσης και προσαρμογής από πλευράς των τριών αυτών μικρών χωρών για να μπορέσει σωστά να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο. Όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Γιατί εδώ μιλάμε για μια συμφωνία σύνθεσης χωρίς ένταξη βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον. Τα φορολογικά μένουν εκτός. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν κάνει αυτές οι τρεις μικρές χώρες υπέρ της διαφάνειας σε δημοσιονομικά ζητήματα και φορολογικά προκειμένου να καταπολεμηθεί η νομοποίηση παράνομου χρήματος και η φοροδιαφυγή. Είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από αυτές τις τρεις χώρες να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον ΩΣΑ, και να ξέρουμε ότι αυτές οι τρεις χώρες είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι στον Κρέκο, είναι στην ομάδα δηλαδή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνουν. Η σύσταση αναφέρει και επιστήνει την προσοχή μας το πόσο σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε τη συνεργασία με τις όμορε χώρες, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία και να φροντίσουμε για καλύτερη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οριζόντια θα υπογραμμίσω τρία σημεία εδώ. Στην περίπτωση τη Ανδόρα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τι προσπάθειε που κάνει στο δημοσιονομικό τομέα. Ιδιαίτερα για τον καπνό, όπου υπάρχει συμφωνία όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την όμορφη χώρα που το ζήτησε, την Ισπανία δηλαδή. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε από πλευρά του Σαν Μαρίνο τι δυσκολίε έχει να εξάγει στις χώρε μέλη εξαιτία τη συμφωνία για το ΦΠΑ και για το Μονακό πρέπει να ξέρουμε ότι έχει πολύ λίγο πληθυσμό αυτόχθονες μονεγάσκους δηλαδή, που είναι μειονότητα στην ίδια του τη χώρα. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ευελιξία, ευθύς ευελιξία, για να μπορέσει η συμφωνία αυτή να εφαρμοστεί με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τώρα θέλω να δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Μίμητσα και να τον παρακαλέσω να τοποθετηθεί. Οι συμφωνίες σύνδεσης με το Ινανδόρα το... και τον Άγιο ε, Μαρίνο και το Μονακό έχουν ενταθεί οι εργασίες. Ε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αυτές έως τον Ιούνιο στιγμή από την οποία θα χρειαστούν ίσως έως και δύο χρόνια ώστε να εγκριθεί το, ο μεγάλος όγκος ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τους εταίρους μας. Όπως ε, ορθά ε, σημειώνει ο κύριος ε, Αγγιλάρ στην έκθεσή του, έχουμε άριστες σχέσεις με τα τρία αυτά μικρά κράτη. Οι τρεις αυτές χώρες είναι περήφανες για την ιστορία τους και για την ανεξαρτησία τους. Και παρόλα αυτά έχουμε τόσα πολλά κοινά. Ανήκουμε όλοι στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια και είναι φυσικό βεβαίω να επιδιώκεται μια ακόμη στενότερη συνεργασία μαζί τους. Εκτιμούμε την επιθυμία τους ε, να ενταχθούν πλήρως στην ενιαία αγορά. Οι τρεις αυτές χώρες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την οικονομική και δημοσιονομική τους ανάκαμψη καθώς και ε, προετοιμασίες για τη μελλοντική συμφωνία σύνδεσης. Για παράδειγμα, έχουν μεταφέρει ήδη στην εθνική ε, ένωμη τάξη τους κάποιους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με το σχέδιο συστάσεών σας, εμείς συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους εταίρους μας να ζητούν την υποστήριξη κατά τη μεταφορά του ευρωπαϊκού κεκτημένου και την υλοποίησή του. Αυτό βεβαίως χρειάζεται, ε, απαιτεί ε, διοικητικέ ικανότητε και εδώ η συνεργασία με τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη. Χαιρετίζουμε το γεγονό ότι στο σχέδιο συστάσεών σα τονίζεται τη σημασία της διατήρησης της, ε, του ενιαίου χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς και του σεβασμού στις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Συμμεριζόμαστε Πλήρω τι απόψει του Κοινοβουλίου και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμία υποχώρηση όσον αφορά τι αρχέ τη εσωτερική αγορά. Αυτέ είναι και οι αρχέ που μα καθοδηγούν στι διαπραγματεύσει μα με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Κάθε συμφωνία θα εμπίπτει εντό των ορίων που θέτουν αυτοί οι κανόνε αυτέ οι αρχέ. Ωστόσο, εντός αυτών των αρχών και κανόνων υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων και διαμισολάβησης που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις που χαρακτηρίζουν αυτούς τους μικρούς εταίρους μας. Και εδώ, σε αυτό το τομέα, είναι πραγματικά επίκαιρες και ευπρόσδεκτε οι συστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει λοιπόν να συνάψει μια ολοκληρωμένη εταιρική συμφωνία που θα καλύπτει και τις τέσσερις ελευθερίες κινήσεων. Η αρχή που μας καθοδηγεί είναι πάντοτε η ίδια ίδια αγορά, ίδιοι κανόνες. Δεν υπάρχει εν μέρη μερική ε, ενσωμάτωση, ένταξη στην ενιαία ούτε μπορεί να προκριθεί η μία ελευθερία έναντι της άλλης. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένου και ενός μηχανισμού ε, για την επίλυση διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί την υλοποίηση και την εφαρμογή της συμφωνίας και στον τομέα των κρατικών επιχορηγήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και με τις αρχές της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσουμε τα αιτήματα αυτών των τριών χωρών για μεταβατική ειδικούς κανόνες ιδίως όσον αφορά την ελευθερία κίνησης εργαζομένων και την ελευθερία παροχή ε, υπηρεσιών και εμπορίες προϊόντων. Οι μεταβατικές αυτές ε, διατάξεις θα πρέπει να είναι αναλογικές. Πάντως, μια συμφωνία σύνδεσης θα είναι αμοιβαία ωφέλιμη, και θα αποτελέσει ένα βήμα για ένα πιο ε, ενωμένο, ε, μια πιο ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Καλησπέρα σε όλους και θα ακούσουμε τώρα τις πολιτικές ομάδες για το ΕΛΚ. Συνάδελφε Ζόφκο, έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Α, δουλεύει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν χαρά για μένα, μη σκιώδη συγγήτρια για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Λόμπε Αγγιγιάρ, για την καθοδήγησή του πάνω σε αυτό το θέμα και του άλλου σκιώδει για επικοδομητική συνεργασία. Σημαντική πτυχή τη εκθέσεω είναι η αναγνώριση τη εδαφική διάσταση αυτών των χωρών και τι συνέπειες έχει αυτό. Μαζί με τους συναδέλφους πρότεινα μέτρα για να θετηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τις τρεις γειτονικέ χώρες να εφαρμόσουν τη μελλοντική συμφωνία σύνδεσης με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Αναμφισβήτητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενθαρρύνει αυτές τις συμφωνίες σύνδεσης με Ανδόρα, Μονακό και Σαν Μαρίνο και τρεις χώρες περιτριγυρίζονται από κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και σαφώ μοιράζονται την ιστορία μα και τι πολιτιστικέ μα αξίε. Αυτέ οι τρει χώρε, η καθεμία από μόνη τη, έχει κάνει σημαντικέ μεταρρυθμίσει και ρυθμιστική ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω σχετικά με τον κανονισμό για τι τράπεζε και τα δημοσιονομικά. Αυτέ οι μεγάλες προσπάθειες θα πρέπει να επενεθούν. Με την οθέτηση τη εκθέσεω. καλούμε για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια απλή συμφωνία, ώστε να βασιστούμε στις μακρά διαρκεία σχέσεις μας με τους γείτονε μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο συνάδελφος Μπονιφέ έχει το λόγο. Παρακαλώ να τον Μπράντο. Εκτό μικροφώνου, ο κ. Μπονεφέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον ηγητή, τον κ. Λόπε, τη Αγγελιάρ. Η συμφωνία σύνδεση μεταξύ Αποξενώσεω, Ανδόρα, Μονακό και Αγίου Μαρίνου είναι σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που σήμερα βλέπει αυτέ τι χώρε να συμμετέχουν που πάντα ήταν ριζωμένε στην ιστορία τη Ευρώπη, αλλά ήταν εκτό του ενωτικού αυτού εγχειρήματο. Για να βελτιώσουμε το κείμενο και για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία, και χάρη στο διάλογο με το κόμμα της πολιτικής μας οικογένειας, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες του Σαν Μαρίνο, ε, υπέβαλα δύο τροπολογίε που έγιναν αποδεκτέ για σημαντικέ πτυχέ, όπω επιστημονική έρευνα και διάδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Τριών Χωρών. Οι διαπραγματεύσει μπορούν να είναι ευκαιρία ώστε να θέσουν πίσουμε μέτρα για υποδομέ, για κοινοφελεί, κοινοφελή θέματα όπω πανεπιστημιακή έρευνα και ανταλλαγέ στον τομέα των επιστημονικών. Θα πρέπει να προλεύουμε και περιοδικέ ακρόσει εθνικών αντιπροσωπιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι θεμελιώδε λοιπόν η ένταξη αυτών τριών χωρών να προχωρήσει αμέσω με τον πιο κατάλληλο τρόπο και για να συζητήσουμε θέματα επί των οποίων μπορούν να υπάρχουν διαφωνίε ή αμοιβαία αιτήματα. Στο σημερινό κόσμο, όσο πιο ενωμένοι είμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο, τόσο πιο ισχυροί είμαστε όλοι μα. Ευχαριστώ για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ο κύριο Τάνοκ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Οι ιστορικές ε, και γεωγραφικές ε, σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά τα τρία μικρά κράτη είναι αδιαμφισβήτητες. Υπάρχει ήδη ένας ικανοποιητικός βαθμός πρακτικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των τριών χρόνων. Και οι τρεις χώρες χρησιμοποιούν το ευρώ, ενώ συμμετέχουν το ο Άγιος Μαρίνος και η Ανδόρα και στην Τελωνιακή Ένωση. 150.000 ε, κατοίκους πληθυσμό έχουν αυτές οι τρεις χώρες μαζί. Γι' αυτό το λόγο η Συμφωνία Σύνδεσης θα αναγνωρίζει αυτή την σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δύο συμβαλόμενων μερών. Και χαίρομαι που η έκθεση Αγγιλάρ ε, τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη της αυτή η διάσταση ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα μικροκράτη στη σύναψη συμφωνιών ε, σύνδεσης. Ε, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πληγεί υπερβολικά ε, η διοίκηση αυτών των χωρών στην, ε, όσον αφορά το καθήκον της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Εγώ ως προερχόμενος από το Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλές φορές αυτές οι τέσσερις ελευθερίες δεν είναι πάντοτε δεδομένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι και προβληματικές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτών των τριών κρατών θα πρέπει να θεωρηθούν κάποιες ε, εξαιρέσεις ε, ως ε, λογικές και να τις χειριστούμε με προτεραιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τον κύριο Αγγιλάρ για την έκθεσή του και θα την υπερψηφίσω αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ συνάδελφε Σολέ για τους πρασίνους. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό είναι τρεις ευρωπαϊκές χώρες με πολύ σαφές ε, κατευθύνσεις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές κλπ. Όπως οι γείτονε χώρες τους, έτσι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας εφέρει να έχουμε πιο στενές σχέσεις και αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης σίγουρα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας. Στις διαπραγματεύσεις που ελπίζω σύντομα να ολοκληρωθούν, να ληφθούν υπόψη οι θέσεις της κοινή γνώμης των τριών αυτών χωρών, που μπορεί κάποιες να είναι επιφυλακτικές για αυτή τη ε, συμφωνία. Εξαρτάται βέβαια από το πώς θα προχωρήσουν και θα, ποιο θα είναι το περιεχόμενο, γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Για την Ανδώρα πρέπει πράγματι να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνει αυτή η χώρα για να αλλάξει τις βάσεις του οικονομικού της συστήματος και επίγει να υπάρχει διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα και να συμμορφώνεται με τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και πρέπει να ζητήσουμε ακριβώς από τις αρχές της χώρας να συνεχίσουν τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τις πολιτικές ομάδες και τώρα μερικές παρεμβάσεις. Ε, συνάδελφε Φίσας, για ένα λεπτό Σαντιάγο, εις το λόγο. Ε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Λόπες Άγκυλαρ, για το έργο του. Είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Πρόκειται μεν για μικρές χώρες, αλλά βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Χαίρομαι όλο ιδιαίτερω για την Ανδώρα, γιατί βρίσκεται κοντά στη χώρα μου και γιατί είμαι και πρόεδρο τη ομάδα φιλία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανδόρας. Η κυβέρνηση της Ανδόρα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά κεκτημένα και προδιαγραφές. Έχουν προχωρήσει από μια σκοτεινή οικονομία σε μια οικονομία ανοιχτή και στον τραπεζικό τομέα και στον τουρισμό. Πρόκειται για μια χώρα πρότυπο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερα υψηλέ προδιαγραφέ ευημερίε. Αυτέ οι τρει χώρε λοιπόν με τα χαρακτηριστικά που έχουν δεν μπορούν μεν να αποτελέσουν μέρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μπορούν να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά μέσω αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριο Άση. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι χώρε, η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιο Μαρίνο αντιπροσωπεύουν πάνω από 115.000 Ευρωπαίου με στενέ ε, σχέσει με τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια έχουν μια πολύ στενά συνδεδεμένη ιστορία με τι ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να νεώσουμε λοιπόν το πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών των χωρών. Και βέβαια πρέπει να πλησιάσουμε αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ε, έναντι της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ακόμα βιώσιμες κοινωνικά και οικονομικά. Αυτή η συμφωνία σύνδεση θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη, αυτή την πρόκληση, να βελτιωθεί η πρόσβαση αυτών των χωρών στην ενιαία αγορά. Αλλά αυτές οι χώρες βέβαια θα πρέπει να καταβάλουν μια προσπάθεια ούτω ώστε να είναι πιο κοντά στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι τράπεζε και τα θέματα διάφορα τη δημοσιονομικά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια εκεί και βέβαια πρόοδο έχει ε, επιτευχθεί μέχρι τώρα. Αυτή η συμφωνία σύνδεση θα πρέπει να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω προτάθηκε, και βεβαίω συμφωνώ ε, με τη δημιουργία μια αντιπροσωπεία ε, διακυμβιστική για διάλογο με τα κοινοβούλια αυτών των χωρών. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τα τρία αυτά μικρά κράτη είναι τα επόμενα. Δεν, δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι τον Πάκμαν που πάει και τρώει τις μικρές τελίτσες. Αν αυτά τα έθνη θεωρούν ότι θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση θα τους παρέπεμπα σε αυτό που είπε ο Επίτροπος. Δεν υπάρχει εν μέρη ένταξη. Υπάρχουν μια σειρά απονομικές πράξει, κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις γύρω από υπαναχωρήσει και προσωρινά opt-out, εξαιρέσει, αναρωτιέμαι πόσο θα διατηρηθούν αυτά πόσο θα γίνονται ανεκτά όσο θα πλησιάζουν οι χώρες αυτές την ε, ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους κανόνες που τις συνοδεύουν. Συμβουλή μου προς αυτές τις τρεις χώρες, σε αυτές τις εξαιρετικές χώρες, θα ήταν προσέχετε, έρχεται ο Πάκμαν, αρχίστε να τρέχετε. Συνάδελφε Τρεμόζα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή Λόπε Άγγελαρ, τους σκιώδη εισηγητέ. και ιδιαίτερα το σατίακοφί σα, γιατί έχουν επιτελέσει εξαιρετικό έργο. Είμαι από τα Πυρηναία, πολύ κοντά στην ε, Ανδόρα. Ιστορικά είχαμε δυσκολίες για χρόνια. Η Ανδόρα τα τελευταία χρόνια πέρασε από μια τεράστια μετάβαση και είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία που ελπίζω να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία αύριο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι όλους αυτούς τους αδέρφου, του οποίους αναφέρθηκα, για τις προσπάθειές τους, για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που βοηθούν την Ανδώρα και όπως είπε και ο συνάδελφο, πρέπει να συγχαρούμε την κυβέρνηση τη Ανδώρα, το κοινοβούλιο τη Ανδώρα και τον πληθυσμό τη το λαό τη, που θέλουν να προσεγγίσουν στις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ο Έχετε το λόγο για ένα μισή λεπτό, για ένα λεπτό μάλλον, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μονακό, η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος είναι τρία μικροκράτη, τα οποία ήταν και είναι γνωστά ως φορολογική παράδειση, ως περιοχές όπου βεβαίως πηγαίνουν πολυεθνικές ή οι πάρα πολύ πλούσιοι και εγκαθίστανται και είναι γνωστός ο ρόλος τον οποίο παίζουν. τώρα με την συμφωνία σύνδεσης υποτίθεται ότι αυτά θα απαλληφθούν. είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος αν αυτό θα συμβεί αν θα σταματήσουν να είναι φορολογική παράδειση αν θα προχωρήσουν με διαφάνεια στις ρυθμίσεις που επιβάλλει η ευρωπαϊκή ένωση. ρωτώ μπορεί κάποιος να ασκήσει δικηγορία στο μονακό; διότι αυτό απαγορεύεται. ρωτώ τι θα γίνει με το οικογενειακό δίκαιο ιδίω στο μονακό που εισάγει διακρίσεις κατά των γυναικών. υπάρχουν θέματα με την επιμέλεια των τέκνων σχέσεις επίσης με τη λειτουργία των τραπεζών. είναι σοβαρά ζητήματα αυτά τα οποία πρέπει να παρακολουθήσει κανείς. ορισμένα από αυτά γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα και γύρω από την έννοια τη ευελιξία δεν πρέπει να επιτρέψουμε όλες αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαρία, ένα λεπτό, τελευταίος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο Φίσας, γιατί πραγματικά έχει δεσμευτεί πάρα πολύ για αυτήν την συμφωνία. Οι τρεις αυτές χώρες συμμερίζονται ιστορία, ενδιαφέροντα και στόχους έχουν τους ίδιους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεωγραφικά ε, είναι βέβαια ευρωπαϊκές χώρες και έχουν υπογράψει και πολλές συμφωνίες μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ανδόρα από το 1990 υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε που συνεχίζει να ισχύει. Ε, πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ και η σύγκληση τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική εναρμόνιση, με την καταπολέμηση ε, του, της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να ενημερωθούν έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν ότι θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία πολύ γρήγορα επειδή η Αμερική προσπαθεί να είναι ηγεμόνα σε, ολόκληρη την, ε, σε ολόκληρο το πλανήτη, είναι καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να επηρεάσει ε, τα πράγματα και θα το κάνει με αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Η έγκριση των συστάσεων ε, θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη και επίκαιρη. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους, για τις προτάσεις τους, για τα σχόλια που έκαναν σήμερα, αλλά και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ στη συνεδρίασή της 21ης Ιανουαρίου. Είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης με τις τρεις αυτές χώρες και για την υποστήριξη που μας παρέσχε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Μίμητσα. Και τώρα θέλω να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι εκπλήσωμε από τη σταθμισμένη αντιμετώπιση η οποία κυριάρχησε στις παρεμβάσεις σήμερα από τις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες. Κάτι το οποίο δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποδεχτεί σε αυτή τη συμφωνία αυτές τις τρεις ε, μικρές χώρες οι οποίες συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ιστορία της. Οπότε θέλω να επιστήσω την προσοχή μας στο ότι εδώ πρόκειται για μια πολιτική δήλωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές τις τρεις μικρές χώρες επικυρώνουμε τη συμφωνία για την σύσταση να προχωρήσει η διαδικασία, για να τη στηρίξουμε, να την προωθήσουμε και να τονίσουμε ότι πρέπει να προχωρήσει με επιτυχία και να σεβαστούμε τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες και στις τρεις περιπτώσεις. Και πρόκειται για μια διαπαιδαγώγηση ουσιαστικά, πρόκειται για τρεις δημοκρατικές χώρες. Άκουσα κάποιες επικρίσεις οι οποίες μπορούν να αναφέρονται κάλλιστα και σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως αυτές οι τρεις χώρες έχουν δεσμευτεί στο δρόμο τον δημοκρατικό. Πρόκειται για μια διαπαιδαγώγηση που κάνουμε, να εξηγήσουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις τρεις μικρές χώρες που δεν ζητούν να ενταχθούν ως μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποψήφιες για συμφωνία σύνδεσης. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε θετικά όσον αφορά αυτή τη συμφωνία σύνδεσης που ελπίζω, ελπίζουμε από ό,τι κατάλαβα να γίνει σύντομα πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν για την εργασία σας. Περατούτε συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Έφτασε ο συγκητής. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση Lockegaard που καταφθάνει με γρήγορο, με γοργό ρυθμό στην Ολομέλεια όσον αφορά τι απαιτήσει προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή. Ορίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι συμβαίνει, το βλέπετε και στο Λονδίνο. Θα είμαι σύντομος. αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί σκιώδεις ηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντική στιγμή αυτή για μας στο Κοινοβούλιο και περίπου για 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι είναι αντικείμενο νομοθεσία θα βελτιώσει προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίε, ούτω ώστε ανεξάρτητα από του περιορισμού ή τυχόν αναπηρίε που έχουν, θα μπορούν να έχουν τηλέφωνο, υπολογιστή ή τηλεόραση που θα είναι προσβάσιμη για αυτούς τους ανθρώπους και θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά όπως κάθε άλλος καταναλωτής. Σε μια κατεπήγωσα ανάγκη μπορείς να, να καλέσεις το 112 για βοήθεια, ε, θα μπορεί να βρει ε, χρόνους, ε, ώρες αναχωρήσεως για κάποια δρομολόγια, να πάρει χρήματα από το αυτόματο μηχάνημα, από το ATM. Για του ανθρώπου χωρί πρόβλημα αυτά είναι απλά πράγματα λέμε. Για ανθρώπου που έχουν περιορισμού, ε, αυτά ήταν δύσκολα. Είναι νομοθεσία που άργησε επί χρόνια και επιβεβαιώνει τι φιλοδοξίε που είχαμε ε, στα πλαίσια τη συμβάσεω του ΟΗΕ για τους ανθρώπου με αναπηρία. Προσωπικά είμαι υπερήφανο για αυτό το κείμενο. Έγιναν σκληρέ διαπραγματεύσει, πήρε πολύ χρόνο, αλλά είμαι υπερήφανο για τα αποτελέσματα που είχαμε. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι το κέντρο για επίγους ανάγκη το 112 θα συμμετέχει τα, τα ATM, ε, μέθοδοι πληρωμής, διάφορες ε, μονάδες ε, παροχής υπηρεσιών για πώληση εισιτηρίων στα τραμ, στα λεωφορεία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Ε, το Κοινοβούλιο μπόρεσε να συμπεριλάβει και τις δημόσιες αγορές μπορέσαμε να, καλύψουμε και πολύ μικρές εταιρείες ε, ε, προβλέπονται κατάλληλες παρεκκλήσεις όταν χρειάζεται. Μιλάμε για λειτουργικότητα και για τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει οι εταιρείε να μπορούν να συμμορφωθούν και να βρουν τις δικές τους τεχνικές ε, λύσεις και προδιαγραφές. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Είναι τα πάντα τέλεια. Όχι. Η αδίποτε διαπραγμάτευση συνεπάγεται συμβιβασμούς. Ε, και είναι κάποιοι που είναι πολύ απογοητευμένοι που δεν συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια. Το ξέρω ότι κάποιοι είχαν ελπίσει ότι θα συμπεριλαμβάναμε περισσότερα και το καταλαβαίνω αυτό σαν εισηγητή. Για να περάσουμε καλά σημεία ε, πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς. Δεν θέλω να τα χάσω όλα. Δεν θέλω να απολεστεί επιτευχθεί σαν πρόοδος για να επιτευχθεί πρόοδος παντού. Ε, προσβλέπω λοιπόν στην αναθεώρηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο χρόνια για να ξέρουμε πόσο προχώρησαν οι διάφορε χώρε. Και ελπίζω να προθεθεί αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κόζα. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό εν ονόματι τη Επιτροπή για Κοινωνικέ Υποθέσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ υπόθηκε και νωρίτερα. Το 2009 ήμουν ο πρώτος ευρωβουλευτής με προβλήματα ακοής, κοφός. Το 2011 εγκρίθηκε το πακέτο για τους ανθρώπους με αναπηρίες, καθώς και η στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, που μας καθοδηγεί στο 2020. Στην έκθεση που είχα συντάξει τότε, είχα ζητήσει από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι με αναπηρίες. Είχα τότε τονίσει ότι σημαντικό στοιχείο είναι η προσβασιμότητα και ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες. Τα τελευταία πέντε χρόνια δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μια ε, νομική πράξη. Όμως, το 2011 η Κομισιόν υπέβαλε μια τέτοια πρόταση και μπορώ να πω ότι ε, μετά από τρία χρόνια διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο είναι θετικό και για τους ανθρώπους με αναπηρία και για τις επιχειρήσεις. Επειδή επίκειται το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας, ήταν ανάγκη να επιταχύνουμε το έργο μας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι συγκινημένος και περήφανος ταυτόχρονα. Εκ μέρους όλων των ανθρώπων με αναπηρίες θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και θέλω να σας παρακαλέσω να βαδίσετε στον ίδιο δρόμο στο μέλλον. Αυτά που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να επιτύχει μέχρι σήμερα θα τα καταφέρουμε στο μέλλον με τη συνεργασία μας. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για όλα όσα έκανε, διότι καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο, το οποίο και θα υπερψηφίσω. Ευχαριστώ, συνάδελφε